χωρίς καθυστέρηση εφόσον ε, είναι παρόν ο εισηγητής θα μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα έκθεση David Martin για την προσαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνθήκη της Λισαβόνας. Κύριε David Martin, έχετε το λόγο. Thank you Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, ανεκτικότητα και την παρουσία σας. Όταν το 2004 έγινε και πρώτη φορά μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είπα στους συνοδέλφους τότε και ειδικότερα στον Κέτ